διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εμπλουτίσει τη σκέψη της και να προωθήσει καλύτερα την κοινωνική αυτή πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση Heinz Karl Becker πρωτοβουλία για τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Τον λόγο και ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Κύριε Μπέκερ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με την ε, πρωτοβουλία αυτή θεωρώ πως κάνουμε κάτι θετικό για την Ευρώπη, ειδικά σε καιρούς δύσκολες, και νομίζω πως δρούμε προληπτικά. Από τη μία έχουμε τις δημογραφικές εξελίξεις και από την άλλη την αγορά εργασίας καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Στην λευκή και στην πράσινη οικονομία, δηλαδή πέραν από τους κλασικούς τομείς οικονομίας που αφορούν ε, την υγεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και το περιβάλλον, προβλέπουμε μία εξέλιξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έναν τρόπο επικοδομητικό και με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές, τη Γραμματεία της Επιτροπής ε, και την Κομισιόν αλλά και τους βοηθούς μου. Το μεγάλο ενδιαφέρον σημείο εδώ πέρα και το μεγάλο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύεται από τις ε, 280 τροπολογίες, 30 συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας στην Επιτροπή μας. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά σημεία εδώ πέρα. Ζητάμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη μελλοντική αυξανόμενη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες με ένα νέο καινοτόμο κλίμα, ειδικά προς συμφέρον των ε, νέων οι οποίοι θα βρουν εδώ πέρα σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Και τι σημαντικότερο υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν πως όλοι πρέπει να ενισχύσουμε αυτές, αυτούς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, ενώσεις, ε, συλλόγους, ε, κοινωνικά ιδρύματα και πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι με ιδιωτικές, με προσωπικές πρωτοβουλίες, ως επιχειρηματίες ή ως ομάδες, ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται, εκμεταλλεύονται τις ε, ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν για να ε, βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτούς τους κοινωνικούς στόχους. Ναι, η έκθεσή μας λέει ξεκάθαρα πως η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι τμήμα της ε, κοινωνικής οικονομίας αγοράς και της εσωτερικής αγοράς, οπότε είναι ισότιμη με όλες τις άλλες μορφές επιχειρηματικότητας. Και εδώ πέρα μία είναι η βασική προϋπόθεση. Το αποδεδειγμένα να έχει κανείς με αυτή την επιχειρηματική του δραστηριότητα μία, ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Είτε μιλάμε για παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, είτε ε, για την φροντίδα ασθενών είτε για τη μετάβαση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Όλα αυτά έχουν σημασία. Η Παγκόσμια Επιχειρηματική Σύνοδος Κοροφής στην ε, Βιέννη έχει προσφέρει χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Ο ορισμός λοιπόν της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αναφέρεται και στο πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού και είναι συμβατός με άλλες εκθέσεις. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αποδειχθεί πως αντέχει στην κρίση. Θέλουμε λοιπόν να την χρηματοδοτήσουμε και περισσότερο στο μέλλον με το ε, κοινωνικό ταμείο το οποίο θα δημιουργήσει και ένα σύστημα σήματοδότησης αλλά και καλύτερη βελτίωση στις δημο... Ε, της πρόσβασης στις δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει επίσης αυτό να ενταχθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ελπίζω στην ανακοίνωση της Κομισιόν να βρούμε κάποια στήριξη. Ελπίζω λοιπόν να ε, υπερψηφιστεί η έκθεσή μου και αύριο στην Ολομέλεια. Υπάρχει εδώ πέρα τεράστιο δυναμικό για να επιλύσουμε κοινωνικά προβλήματα και έτσι η Ευρώπη να αποτελέσει κοινωνικό πρότυπο στον κόσμο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν το 10% όλων των ευρωπαϊκών εταιριών και απασχολούν ε, ε, ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να ε, σχετίζεται και με την βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο με επιδοτήσεις, γιατί μόλις λήξει η επιχορήγηση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ε, σκεφτόμαστε ότι η οικονομική υποστήριξη θα πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση της απόσβεσης που θα έχει η επένδυση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται από αυτούς τους ε, μηχανισμούς χρηματοδότησης. Και είναι πολύ δύσκολο να βρουν αυτές τις πληροφορίες. Χρειάζεται μια, ε, χρειάζονται σαφέστεροι και απλούστεροι κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μπέκερ για τη δουλειά που έκανε για αυτήν την έκθεση και για την συνεργασία του με όλους τους σκιώδεις συγητές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβαλούν σε μεγάλο βαθμό στην απασχόληση, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία και τα μειονεκτούντα άτομα. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πραγματικές επιχειρήσεις. Πραγματοποιούν κέρδη και τα επενδύουν. Θα ε, ε, ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να μειώσουμε το διοικητικό άκθος για τις ε, επιχειρήσεις αυτές όπως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει ένα παράδειγμα μια λατινικής επιχείρησης που απασχολεί άτομα με αναπηρίες, ανταγωνίζεται στην ανοιχτή αγορά και το επιτυγχάνει. Ανήκει ε, σε, μια, σε ένα ευρύτερο δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ονομάζεται ε, Mobilis και που ε, αξίζουν όλη την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινωνική οικονομία έχει υψηλή ικανότητα αντοχής στην κρίση και αλληλεγγύη και, έχει ε, μια ε, ε, μεγάλη ανθεκτικότητα. η υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών έχει κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων ευνοεί την δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δημοκρατικής, πιο συνεκτικής, πιο αλληλέγγυας, που είναι ικανή να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η βελτίωση λοιπόν του νομικού και φορολογικού πλαισίου είναι κάτι που απαιτείται και μια ε, οικονομική υποστήριξη από την ε, Ευρώπη, ε, πιο ευνοϊκή μεταχείριση και πρόσβαση στα δημόσια έργα που θα μπορούσε να ευνοήσει την οικονομική αλληλεγγύη και η οικονομική, με συγχωρείτε, ανεξαρτησία των επιχειρήσεων αυτών για τη δημιουργία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό ευχαριστώ τον συνάδελφο για την δουλειά του. Κυρία Τικάου είναι ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο κοινωνικών επιχειρήσεων είναι σημαντικέ παρά το γεγονό ότι οι κοινωνικέ επιχειρήσει καλύπτουν το 10% τη απασχόληση. Εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο οι επιχειρήσει αυτέ για να μπορέσουμε να έχουν το ρόλο τους. Αυτό όμως απαιτεί μια χρηματοδότηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι μέσω του Κοινωνικού και του Περιφερειακού Ταμείου θα έχουν καλύτερη χρηματοδότηση και θα έχουν και την απαραίτητη ευκαμψία τα κράτη-μέλη προς το σκοπό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε το πνεύμα του επιχειρήν να έχουμε καινοτόμε επιχειρήσει κοινωνικού χαρακτήρα που να κατευθύνονται περισσότερο προ του νέου και τα άτομα με μειονεξίε. <clears throat> θα πρέπει να συνεχίσουμε <clears throat> το πρόγραμμα Εράσμου για του νέου επιχειρηματίες και να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνική οικονομία. Και η κυρία Μπασέσκου είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ την συνάδελφό μου για το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρας στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ανάγκη κοινωνικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των δημογραφικών αλλαγών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο μέσα στα πλαίσια αυτά. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να έχουν ένα γενικό ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε, οικονομή, σε ιδιωτική ε, χρηματοδότηση και να κινητοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προστατεύουν να δώσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση με μια τροποποίηση <clears throat> τη ένωμη τάξη τη, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα σε δημόσια χρηματοδότηση αυτή η φορή. Και επίση να βελτιώσουμε τι δυνατότητε διαχείριση από τι κοινωνικέ επιχειρήσει. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν μέσω προγραμμάτων όπω είναι ο έρασμο για του νέου επιχειρηματίε. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. κύριος Ματούλα έχει το λόγο. είναι ανάγκη να είναι κανείς επίμονος και φιλόδοξος σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Χρειαζόμαστε οραματίστριες εταιρείες που να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κοινωνικού συστήματος για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλοι το κέρδος που έχουμε όλοι από τις κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις και να δώσουμε προτιμησιακά υπό χρηματοδότηση σε αυτές τις επιχειρήσεις αντί να έχουμε προγράμματα κοινωνικής, κοινωνικών παροχών. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα που θέλει να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία και του δημόσιου τομέα και να δω, που θέλει να δώσει κοινωνική υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα χρήματά μας και να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι κοινωνίες, επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να υποστηριχθούν από, τις, ε, από τα κοινοτικά ταμεία και να πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε πολλαπλά τέτοια ταμεία και να τύχουν και τη υποστήριξη των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη προώθησή του, ώστε να μιμοποιηθούν και οι πρωτοβουλίε που κάνουν αυτέ οι επιχειρήσει. Ευχαριστώ. And next Ευχαριστούμε, κυρία Ρέγνερ. Κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν και ιδιαίτερα εσείς, Επίτροπε Μπαρνιέ, αναλάβατε μεγάλες δεσμεύσει και πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και το καλωσορίζουμε. Υπάρχει όμως ένα θέμα που θέλω να θέσω σε σχέση με την πρόταση αυτή για την κοινωνική οικονομία. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα πρέπει να ανοίξει, ε, αλλά αυτό δεν έχει γίνει σωστά θα πρέπει οι επιχειρηματίες να δεσμεύονται υπέρ κοινωνικών στόχων και επανεπένδυσης. Αυτό το ταμείο δεν είναι το καλύτερο. Ήδη υπάρχουν αρκετές δυνατότητες όπως ε, ε, αναπτυξιακές τράπεζες, ε, συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα πρέπει να οργανώνεται με τρόπο δημοκρατικό και αλληλέγγυο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόγαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, όμως υπάρχει μια επαρκής χρηματοδότηση, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε περαιτέρω χρηματοδοτικά μέσα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια λύση θα μπορούσε να, να την, πρόσθεση, την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία που είναι σχετικά δηλαδή τα διαφορετικά ταμεία που χρηματοδοτούνται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης μια άλλη λύση θα ήταν να έχουμε τον ορίζοντα 2020, το σχετικό ταμείο, το πρόγραμμα για τις κοινωνικές αλλαγές και την καινοτομία και επίσης πρόσβαση για μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μόνο έτσι δεν μπορούσαμε να δώσουμε επαρκή υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις που προωθούν εργα... θέσεις εργασίας υψηλού επίπεδου, καταπολεμούν την ανέχεια και την... τον κοινωνικό αποκλεισμό και επενδύουν στην επαγγελματική μετάρρυνση των Ευρωπαίων. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κ. Σογκόρ. Ευχαριστώ. Σε αυτό το διάστημα που επίκειται, η οικονομική κρίση θα δείξει πολλές επιπτώσεις. Πιστεύουμε όλο και περισσότερο ότι στα πλαίσια της καταπολέμησης της κρίσης είναι πολύ σημαντική η αντιμετώπιση του χρέους. Όμως Λίγα μένουν, ε, ε, ε, λίγο ασχοληθήκαμε με τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Διατυπώθηκαν διάφορες προϋποθέσεις. Οι πολίτες όμως έχουν την αίσθηση ότι δεν ασχοληθήκαμε αρκετά με την αυξανόμενη ανεργία, τα κοινωνικά προβλήματα, τη φτώχεια. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ξέρουν πολύ καλά ποιες επιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν αν παραγνωρίσουμε κάποια κοινωνικά θέματα. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως και σε πολιτικό επίπεδο να ρυθμίσουμε τα κοινωνικά θέματα με κοινέ προσπάθειες, με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιτρέπεται τα ευρωπαϊκά κράτη να θυσιάσουν τα κοινωνικά συστήματα λόγω των επιπτώσεων της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους εσάς και τον κύριο Μπέκερ ειδικότερα και όλους τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντες σε αυτή τη συζήτηση με ένα σημαντικό κατά την άποψή μου θέμα πάνω στο οποίο εργαστήκαμε πολύ εδώ και μήνες με τον συνάδελφο Ταλιάνη για να χαράξουμε αυτό το φύλλο πορείας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα όλες αυτές οι επιχειρήσεις ε, έχουν διαφορετικό καθεστώς στα 27 κράτη-μέλη μας και καλύπτουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και επίσης συμμετέχουν σε σημαντικές επενδύσεις. Αυτά που μας είπε ο κύριος Μπέκερ είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι στηρίζουν την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει μέσα από μια σειρά πρωτοβουλειών και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και με την ίδια επιμονή πρώτον σε ό,τι αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, διότι τον Οκτώβριο 2011 προτείναμε οι κοινωνικές επιχειρήσεις της αλληλέγγυας οικονομίας να αποτελέσουν αντικείμενο προτερότητας για τη χρηματοδότηση με τη νέα γενιά των, των ταμείων μέχρι το 2020. Αυτή είναι μια πρόταση βεβαίω τη Επιτροπή, η οποία θα χρειαστεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Είμαι επίση ευτυχή που διαπιστώνω ότι η ένταξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από την πρόταση για του προγράμματο για τι κοινωνικέ αλλαγέ και μεταρρυθμίσει ε, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία τον περασμένο μήνα. Επίσης οργανώσαμε το πακέτο για τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος προβάλλοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις όταν παρέχουν κοινωνική υπηρεσία. Τώρα, για την ιδιωτική χρηματοδότηση με την έκθεση του ο κύριος Μπέκερ υποστηρίζει ένα σχέδιο κανονισμού για ένα ταμείο επιχειρη... κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχει προτείνει το... Ε, ο... άλλωστε η Επιτροπή. Μιλάμε για ε, ιδιωτικά ε, κονδύλια. Ο σκοπός δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε κρατικά κονδύλια. Όταν υπάρχουν ιδιώτες επενδυτές και θέλουν αυτοί να επενδύσουν σε έναν τομέα ε, όπως οι νέες επιχειρήσεις Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια διευκόλυνσης και προώθησης αυτής της χρηματοδότησης με αλληλέγγυο τρόπο και αυτό δεν αντιβαίνει καθόλου με άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες κινητοποιούν και κάνουν χρήση δημόσιων κρατικών κονδυλίων. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το Ταμείο ε, κοινωνικής, ε, κοινωνικής ε, Επιχειρηματικότητας και ότι θα, θα, θα αυτή η προσπάθεια με επιτυχία. Και για τους φορολογικούς παράδεισους πρέπει να, νομίζω να καταλήξουμε σε μια δυναμική συμβαστική λύση. Τώρα πέρα από τα οικονομικά θέματα γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ε, θέλει να προωθήσει την ε, ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ήδη στην πρόταση του 2000 ε, η σχετική πρόταση της Επιτροπής πριν από λίγα χρόνια δεν είχε γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και αποσύρθηκε. Υπάρχει και το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε ε, σχετικά με αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει πρόοδος. Συνάντησα σημαντικά στελέχη των ε, ε, ιδρυμάτων που υποστηρίζουν, που υποστηρίζουν την πρότασή μας. Επίσης, για τις ε, δημόσιες συμβάσεις και αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα εφόσον υπάρξουν κανόνες που θα ε, συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη, στην προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Ε, ε, έχουμε προχωρήσει σημαντικά στη δουλειά που έχουμε κάνει για να υποβάλουμε τις προτάσεις το οι οποίες θα σας υποβληθούν σύντομα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις πρωτοβουλίες μας, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε και σε συνεργασία με τον κύριο Τελιάνη και τον κύριο Ντόρ θέλουμε το Single Market 2, η ενιαία πράξη 2, ε, να αποτελέσει ένα μοχλό για την προστασία των καταναλωτών, για την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στα πλαίσια ε, αυτής της ε, πράξης θα προωθήσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα, θα προσδιορίσουμε τι είναι ακριβώς μέσα στην ποικιλομορφία τους οι κοινωνικές επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε την αξιοπιστία τους έναντι των επενδυτών, κάτι που υπογραμμίζει επίσης την έκθεσή του ο κύριος Μπέγκερ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο διευκόλυνσης που θα συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών βέλτιστων πρακτικών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπως το έχετε ζητήσει, εγγραφή στα πανεπιστημιακά προγράμματα, το έρασμος, και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είμαστε μόνοι, δεν ενεργούμε μόνοι και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρέπει να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, ένα βήμα ανταλλαγών. Ξεκινήσαμε με μια σημαντική διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν τον Νοέμβριο του 2011 πολλοί από εσά. Ο κύριος Μπέκερ είχε την ευκαιρία τον περασμένο Ιούνιο να ανταλλάξει ε, ε, απόψεις με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή συνοδεύεται ε, από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και αρχές του 2014 θα οργανώσουμε πάλι μια μεγάλη συνάντηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα για να δούμε τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια και να προβλέψουμε και να ε, οργανώσουμε νέες δραστηριότητες για το μέλλον. Στις αρχές του 2014, όπως σας είπα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα, στην